και συνεχίζουμε με το προσεχές θέμα στην ημερήσια διάταξη και γυρνάω πάλι στα γερμανικά. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι προφορικές ερωτήσεις ε, για απάντηση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την ανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κλοντ Μωράης είναι ο πρώτος ο συντάκτης που λαμβάνει το λόγο. Περιμένω ε, έως ότου καθίσει ο Επίτροπος. Θα ήθελα να τον ε, καλωσορίσω καταρχήν, γιατί θα ήταν αγενές να μην το κάνω. Νομίζω ότι όλοι στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θεωρούμε ειλικρινά ότι θα, θέλουμε, θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας εδώ τα καταφέρνουμε καλύτερα. Να προστατεύουμε τους πολίτες μέσα στα πλαίσια μιας προστιθέμενης αξίας. Αυτό είναι ένας δυναμικός και ενδιαφέρον τομέας. Έχουμε να κάνουμε με μια τάμπουλα ράζα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουμε αντιμετωπίζουμε έναν ευαίσθητο τομέα. Υπάρχει τρομοκρατία μέσω ε, κυβερνοχώρου, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και νομίζω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με βάση την εμπειρία και πείρα μας θα θέλαμε να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα αρμοδιότητας του Συμβουλίου αλλά μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς ιδιαίτερα στην εξισορρόπηση μεταξύ προστασίας πολιτών, βεβαίως εγκυόμενη και την διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη. Η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και τις ε, διασυνοριακές ε, ρήξεις και σειράξεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ξένους μαχητές οι οποίοι προσχώρησαν σε ακραία κινήματα και μετά επιστρέφουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτή την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας με βάση την πολιτική της Επιτροπής που θα οριστεί του χρόνου. Θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία αυτός ο τομέας για να βελτιώσουμε τη στρατηγική. Με αυτό το ψήφισμα καθιστούμε σαφές από πλευράς Κοινοβουλίου του τι θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Δεν θέλουμε να, παρά να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και να μπορέσουμε να ε, έχουμε μία ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές. Ιδιαίτερα μας απασχολεί το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και θεωρώ ότι θα πρέπει να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές όπως κάνει το ψήφισμα και να δούμε ποια είναι τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτή την στρατηγική. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας καλύτερα πριν δημιουργήσουμε καινούρια. Αυτό ακριβώς ε, λέμε στο ψήφισμά μας. Θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε τα μέσα αυτά σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο να αντλήσουμε από τα διδάγματα αυτά πριν προχωρήσουμε σε νέα μέσα. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, να χρησιμοποιήσουμε τα προϋπάρχοντα μέσα όπως κοινέ ομάδες, εξεταστικές ομάδες ή έρευνας όπως ορίσαμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα πρέπει να έχουμε εξισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτό το είδαμε από την προστασία δεδομένων, από την εποπτεία του χώρου, του διεθνούς χώρου και όλα αυτά συμβαδίζουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα από πλευρά Κοινοβουλίου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις απειλές στον κυβερνοχώρο, λαμβάνοντας υπόψη πολυσχηδή ζητήματα σε σχέση με τους ξένους μαχητές, την προστασία προσωπικών δεδομένων επιβατών και ούτω καθεξής. Έχουμε πείρα και στον τομέα ασφάλειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι το 2015 θα πρέπει να αντιδράσουμε με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής ως Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, δώσει τη θέμενη αξία έναντι των θέσεων του Συμβουλίου. Εμείς θα συνεισφέρουμε σε αυτή την στρατηγική, έχουμε πείρα και θα ήθελα να ακούσω και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που θα σας δώσουν το κατάλληλο input τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μωράης. Εξ του Συμβουλίου το ε, λόγο έχει ο κύριος Ντελαβέντοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανανέωση της ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Είναι ένα κατά προτεραιότητα θέμα της Προεδρίας. Γι' αυτό χαίρομαι διότι μου δίνετε την ευκαιρία να σκιαγραφίσω τις βασικές μας προτεραιότητες της ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Καταβάλλονται προσπάθειες για να δοθεί συνέχεια στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου για να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια κατά το πρώτο εξάμεινο του 2015. Άρχισαν λοιπόν οι συζητήσεις των Υπουργών τον Ιούνιο για να συνεισφέρουμε στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα ανανεώσει την ανακοίνωσή της την Άνοιξη φτάσαμε σε μία συμφωνία σε σχέση με την ανανέωση της στρατηγικής που αφορούν την γενική διάρθρωση όπως και ορισμένες θεμελιώδεις πτυχές που σχετίζονται και απαντούν στο ερώτημα η ανανεωμένη αυτή στρατηγική θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας ε, τα τελευταία χρόνια. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα σε όλες τις εκφάνσεις του, είτε πρόκειται για τορμοκρατία ή εγκληματικές ενέργειες και χρηματοδότηση του εγκλήματο. Το θέμα των ξένων μαχητών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα όταν επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης γιατί αυτό αποτελεί σημαντική απειλή χωρίς προηγούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο αναγνώρισε και απειλές στον κυβερνοχώρο με βάση τη χρήση νέων τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές καταστροφές ή τις καταστροφές που προέρχονται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ευρύ φάσμα μέσων μέσα στα πλαίσια και της λήψης αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο μέχρι το ευρωπαϊκό και διεθνές. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι ολιστική και να σχετίζεται με πληροφορίες και κατασκοπία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το, τη διεθνή, και το διεθνές έγκλημα, στο οποίο θα προσδώσουμε μεγάλη σημασία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, ο τομέας της δικαιοσύνης είναι ύψης της ε, σημασίας τα δικαιοδοτικά μέσα θα πρέπει να βελτιωθούν και φυσικά θα πρέπει να κατάσχονται τα έσοδα που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ε, ένα καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης ε, των δικαστικών αποφάσεων. Θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση των συνόρων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες εχμής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. το θέμα των ξένων μαχητών δείχνει πτυχές ε, της εξωτερικής και εσωτερικής συνεργασίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύσουμε τους πολίτες μέσα στα πλαίσια της στήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα όσων επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, η ανανεωμένη στρατηγική θα πρέπει να εφαρμόσει όλα τα νομοθετικά μέσα. Το Συμβούλιο πρώτα την, ε, ε, η Επιτροπή να υποβάλει μια ετήσια έκθεση για τη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να εποπτεύσουμε τις εξελίξεις και να μας ενημερώνει η Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις ως προς το χρονοδιάγραμμα της νέας στρατηγικής θα πρέπει να δούμε πώς θα ληφθεί η υπόψη από το Συμβούλιο και η συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Για την ανανέωση λοιπόν αυτής της στρατηγικής ορίζουμε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Όλα εξαρτώνται βεβαίως από την ανακοίνωση της Επιτροπής. Θεωρούμε όμως ότι θα είναι διαθέσιμη κατά την Άνοιξη. Άρα θα μπορέσει να επέλθει συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Όπως ξέρετε, η Προεδρία μαζί με την Επιτροπή διοργάνωσε μία διάσκεψη υψηλού επίπεδου το Σεπτέμβριο του 2014. Ο κύριος Μωράης ήταν ο κύριος ομιλητής. Έτσι συνεισέφερε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό κείμενο του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και την τελική έκθεση της Επιτροπής, η οποία λάμβανε υπόψη και το δικό σας ψήφισμα. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συνεισέφερε πολύ. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι περιμένω με ενδιαφέρον τη δική σας συνεισφορά και είμαι σίγουρος ότι οι συστάσεις σας θα είναι πολύτιμες και θα ενταχθούν στην ανανεωμένη στρατηγική για να γίνει καλύτερη χρήση των ε, υπαρχόντων μέσων πριν δημιουργήσουμε νέα, για να υπάρχει μία σφαιρική προσέγγιση και καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Αναφερθήκατε και στη σημασία του δικαστικού τομέα. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής λοιπόν δημοκρατικός έλεγχος από όλες Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντελαβέντοβα και θα ήθελα ο κύριος Αβραμόπουλος να λάβει το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Αυτή η προφορική ερώτηση λαμβάνει χώρα υπό τη σκιά ενός αποτρόπαιου εγκλήματος το οποίο συνέβη σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου και τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια αθών ζωών σήμερα στο Πακιστάν. Σε ένα πολιτισμένο κόσμο τέτοιου είδους βίες ε, επιθέσεις όπως αυτή που έλαβε χώρα σήμερα σε ένα σχολείο στο Πακιστάν αποτελούν προσβολή για την ανθρωπότητα και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και σε ό,τι θεωρούν ιερό όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό το τραγικό γεγονός και αυτή η αδυσόπιτη δολοφονία μικρών παιδιών δείχνουν πόσο αποτρόπαιο είναι το πρόσωπο των τρομοκρατών. Η τρομοκρατία αποτελεί μια παγκόσμια απειλή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συστρατευτεί για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους συνεργάτες μας για να προστατεύσουμε το δικαίωμα στη ζωή όλων ανεξάρτητα από φιλή, εθνική καταγωγή ή ε, θρησκεία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αγαπητοί ευρωβουλευτές που μου δώσατε την ευκαιρία σήμερα να σκεφτούμε μαζί ποια θα είναι η ανανεωμένη εσωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ασφάλειας αυτή η νέα λοιπόν, το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να είναι κοινό πρόγραμμα όταν η ασφάλεια των συμπολιτών μας, τα δικαιώματά τους, οι δημοκρατικές τους αξίες, η ευημερία της κοινωνίας μας και των οικονομιών μας διακυβεύονται. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν στενά. Χρειάζεται να βρούμε τον κοινό τόπο να βρούμε ποιες είναι οι βασικές αρχές, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες έτσι ώστε να ανανεώσουμε αυτή την εσωτερική πολιτική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως όλα τα θεσμικά όρονα θα πρέπει να συνεργαστούν για να διατυπώσουν και μετά να εφαρμόσουν την μελλοντική ατζέντα της Ευρώπης για την ασφάλεια και να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία. Εάν εξετάσουμε ποια είναι η στρατηγική αυτή τη στιγμή, θα βρούμε διάφορα στοιχεία από τον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε, γιατί έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ήδη και εργασία προετοιμασίας φέτος. Έχουμε τα συμπεράσματα ΔΕΗ που εγκρίνθηκαν στην, την 5η Δεκεμβρίου. Έχουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που θα εγκριθεί που σκοπεύει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο αύριο. Οι συνεισφορές αυτές θα μας καθοδηγήσουν στις εργασίες μας τους επόμενους μήνες. Προτείνω λοιπόν, αφού η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιαστεί, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν ένα διάλογο για να βρουν ε, το κοινό τόμο που θα μας επιτρέψει να έχουμε αποδοτική, γρήγορη εύχρηστη, βιώσιμη ευρωπαϊκή εσωτερική ασφάλεια. Το δικό σας ψήφισμα ακολουθεί μια γενική ευρεία προσέγγιση που βασίζεται σε κάποιες αρχές και δεν απαριθμεί συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις και πολιτικές. Αυτό αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες που έχει εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει μια, ένα πρόγραμμα ε, που θα ε, απορρέει από ε, τις προτεραιότητές μας και που ήδη συμπεριλαμβάνει κάποια φιλόδοξα μέτρα. Το ψήφισμα τονίζει επίσης το πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ συνέχειας αλλά και αλλαγής. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα οποία λειτουργούν και να προσαρμόσουμε ε, τα σημεία στα οποία οι εξελίξεις τρέχουν, όπου χρειάζεται νέα δράση, όπου πρέπει να αναθεωρήσουμε δράσεις του παρελθόντος. Η εφαρμογή της νομοθεσίας και η παγίωση των επιτυχιών μας όπως επίσης και η ενισχυμένη ε, συνεργασία στην πράξη θα αποτελέσουν τις προτεραιότητες για τις μελλοντικές μας εργασίες. Ακολούθως μια παρακολούθηση και μια αξιολόγηση της ε, αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας μας. Και αυτό είναι ουσιαστικό. Το Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε η εποχή κατά την οποία τα θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης ε, βρίσκονται πια σε ισότιμη σχέση με άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη στην πλήρη εφαρμογή της δικαστικής αναθεώρησης που έκανε το ΔΕΚ και των ε, νέων ε, αρμοδιοτήτων, εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται λοιπόν μια αξιολόγηση που θα ενισχύσει τη νομική βεβαιότητα αλλά και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Η στενή παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων υιοθετημένων ε, των νέων εργαλείων για τα δικονομικά δικαιώματα για παράδειγμα και η βελτίωση της ε, νομοθεσίας για τη συνεργασία, για τη δικαστική συνεργασία ε, σε θέματα ποινικά ε, είναι σημεία στα οποία στέκεται και το δικό σας ψηφίσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τακτικές εκθέσεις για τις δράσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για θέματα ασφαλείας. Αυτό θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε το, την εφαρμογή της στρατηγικής και θα ενισχύσει ε, την δημοκρατική εποπτεία σε αυτά τα θέματα. Σε σχέση με το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για την Ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μπει σε λεπτομέρειες για τα θέματα στα οποία, ε, τα οποία θα εντάξει στην ε, μελλοντική της ανακοίνωση. Αναμφίβολα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες πάταξης διεθνούς και διασυνοριακού εγκλήματος, πρόληψης τρομοκρατίας, αντιμετώπισης της ε, ζωστικοποίηση ε, των εξτρεμιστών να βοηθήσουμε να μην υπάρχει ε, καμία εκμετάλλευση παιδιών και να οικοδομήσουμε το χώρο δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Τίποτα καινούριο. Αυτό που είναι η καινοτομία μας είναι πως οι νέες αυτές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν μεταλλασσόμενο κόσμο και απειλές που συνέχεια εξελίσσονται. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση λοιπόν για να δούμε πώς μπορούμε γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προκλήσεις. Ανάλυση απειλών μέσω της ε, Europol για παράδειγμα και άλλων ε, ευρωπαϊκών θεσμών και φορέων σε στενή συνεργασία έτσι ώστε να είμαστε πιο επιχειρησιακοί στην προσέγγιση που ακολουθούμε. Αυτό τι απαιτεί. Στρατηγική και πολιτική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, διοκτικών αρχών και των ευρωπαϊκών φορέων και υπηρεσιών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά για να προλάβουμε και για να προστατεύσουμε. Πρόσβαση στις πληροφορίες, ανταλλαγή πληροφοριών, καινοτομία, έρευνα. Όλα αυτά σε στενή συνάρτηση ε, με την εξωτερική διάσταση της συνεργασίας. Ε, να στοχεύσουμε ε, στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και μία από τις βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική εσωτερικής ασφάλειας. Θα παρακολουθήσουμε στενά το πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα προτινόμενα μέτρα και εργαλεία και θα αξιολογήσουμε ε, την αποτελεσματικότητά τους όπως και πώς επηρεάζουν την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μέτρα, αν χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία ε, επηρεάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να γίνει αυτό με έναν ανάλογο τρόπο έτσι ώστε η πρόληψη κάποιων δημοσίων κινδύνων ε, να νομιμοποιούν αυτή την πίεση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η έλλειψη αυτής θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Οι πολιτικές ασφάλειες θα πρέπει να ε, στηρίζονται και να νομιμοποιούνται από τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και η εφαρμογή της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας δεν είναι μόνο ουσιαστική για να είναι αποτελεσματικά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, αλλά επίσης για να ενισχύσει ε, την αξιοπιστία που έχουν ε, τα ε, ευρωπαϊκά όργανα στα ε, μάτια των πολιτών. Για να εξασφαλίσουμε πως η εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει δράση και εκτός των συνόρων μας και σε συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση των βημάτων που έχουν γίνει στα εξωτερικά και στα εσωτερικά ε, σύνορα. Για παράδειγμα, κυβέρνο ασφάλεια. Ένα παράδειγμα σας έδωσα, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα και ακόμα πάρα πολλά ε, χρειάζεται να δρομολογήσουμε. Για παράδειγμα, ε, μεγαλύτερη διασύνδεση πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θέλετε ένα ολοκληρωμένο, ε, ολοκληρωμένο με ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση στις διάφορες αυτές πολιτικές, γιατί υπάρχουν δράσεις οι οποίες ε, ξεφεύγουν από τα στενά χωράφια αυτής της πολιτικής, ε, γιατί ξέρετε ότι σε πάρα πολλούς χώρους έχουμε ανησυχίες, έχουμε και δημοσιονομικές πιέσεις είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, και το πλεονέκτημα που προσφέρει η έρευνα, η τεχνολογία. Να κινητοποιήσουμε τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να είμαστε πάντα έτοιμοι για να δώσουμε μια απόκριση. Ε, χρειαζόμαστε τις τεχνολογίες πληροφορικής, ε, όπως επίσης και κάποιες προθυμένες τεχνολογίες εγκληματολογικές. Χρειάζομαστε καινοτομία και έρευνα. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω του Horizon 2020. Έτσι ώστε ο ιδιωτικό κλάδος και οι ιδιωτικέ αρχέ να συνεργαστούν όχι μόνο για να προωθήσουν και ε, τεχνολογία εχμής αλλά και για άλλους λόγους. Θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα στα μάτια του Ευρωπαίου πολέτου, ε, πολίτη με μέσω της απόλυτης εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκτός από τις επίσημες εκθέσεις για την εφαρμογή των στρατηγικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμηση να κάνει συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συζητεί τα θέματα αυτά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Προσμένω λοιπόν στη συνεργασία με εσά και με το Συμβούλιο για αυτό το νέο ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα, τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την εσωτερική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, θα ήθελα η κυρία Χολμάιερ να λάβει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ε, ε, κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φυπουργέ, αγαπητοί συναδελφοί, οι διεθνείς ασφάλεια, η στρατηγική μας και οι απαντήσεις που θα δώσουμε στο ζήτημα της ασφάλειάς μας τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκες. Στην τελευταία θητεία είχαμε μάλιστα μία επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη λεγόμενη ΚΡΙΜ, επιτροπή Κρίμα, που είχε σαν στόχο να μελετήσει το οργανωμένο έγκλημα και την παγκόσμια διαπλοκή του. Είναι συγκλονιστικό το να βλέπουμε το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, τις σχέσεις μεταξύ των ε, τρομοκρατιών και των εξτρεμιστών που σήμερα τόσο κατάφορα είδαμε να φωνεύουν αθώα παιδιά. Είδαμε οργανωμένα δίκτυα που εγκληματιών που καθιστούν ε, την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα παιχνίδι για παιδιά εάν δούμε τι πραγματικά εγκλήματα διαπράττουν. Όπω είπε ο κύριο Κλοντ Μωράη, πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη θυσή μα. Όταν η δικαστική αρρωγή κρατάει μήνε για να παρασχεθούν οι πληροφορίε που χρειάζονται ή να ε, υλοποιηθούν τα αιτήματα των δικαστικών αρχών, έχουν πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμαστούν και να διαφύγουν οι εγκληματίε. Χρειάζεται βεβαίω και η προστασία των προσωπικών δεδομένων να εξασφαλιστεί επί πιο καλό τρόπο. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάτη, για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να πω ότι έχει μεγάλη σημασία και δεν πέφτει στο κενό, έρχεται την κατάλληλη στιγμή αυτό το ερώτημα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι προκλήσεις ασφάλειας που έχουν αλλάξει άρδιν τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την ανησυχητική ε, συνάρτηση των νέων απειλών στον ε, κυβερνοχώρο από το διεθνές έγκλημα και την ε, τρομοκρατία. Ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη το διασυνοριακό έγκλημα και τη, την πρόσμιξη αυτή απειλών που σχετίζονται πολλές φορές και με φυσικές καταστροφές. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προστιθέμενη αξία στον ορισμό και την ανταπόκριση μέσα στα πλαίσια της ανανέωσης αυτής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για το 15 έως το 19. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη έχει αλλάξει δραστικά και θα πρέπει να βελτιώσουμε τα μέσα μας, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, συνεργασία της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και της ανταλλαγής πληροφοριών μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με βάση τις αξίες μας, δηλαδή ε, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει μία συνοχή και συνέπεια για την προστασία δεδομένων και για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ερμηνεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό η στρατηγική μας θα πρέπει να τηρεί απόλυτα το, τα πολιτιστικά δεδομένα των, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η κυρία Βονστόρκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα στην, στην ημερήσια διάταξη και το ψήφισμα συζητούμε την εσωτερική ασφάλεια. Και σαφές είναι το εξής, ότι η κατάσταση της ασφάλειας στην Ευρώπη έχει ριζικά αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Στη Γερμανία είναι πολύ επίκαιρο θέμα, είναι το υπαριθμόν ένα θέμα, γιατί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται πια ασφαλείς. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ε, τους, έχει εγκαταλείψει η πολιτική και δεν διασκεδάζει τους φόβους τους. Γι' αυτό και κατά χιλιάδες κατεβαίνουν κάθε Δευτέρα στους δρόμους οι άνθρωποι στη Γερμανία και κάθε Δευτέρα είναι όλο και πιο πολύ. Πρέπει λοιπόν να δώσει απαντήσεις η πολιτική και όχι να δυσφημεί και να καθυβρίζει αυτούς που κατεβαίνουν στον δρόμο. Πρέπει να κάτσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Και πρέπει να δούμε αν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε ανοιχτά για τα προβλήματα να αναγνωρίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και μόνο έτσι μπορούμε να το λύσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μλίναρ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Ντελαβέντοβα, στη Λίμπε φτάσαμε σε ένα συμβασμό μεταξύ πολλών πολιτικών ομάδων και ελπίζω να λάβετε υπόψη τις σκέψεις μας κατά την ανανέωση της στρατηγικής. Με βάση την προηγούμενη στρατηγική, δηλαδή μάλλον μετά την έγκριση της προηγούμενης στρατηγικής, ήρθε ετέθη σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική της αποτίμηση. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μία συμφωνία ε, επί της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων για λόγους ένομης τάξης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία ύψης της σημασίας μέσα στα πλαίσια του πολιετούς ε, πλαισίου. Θα ήθελα να υποστήριξουμε το κείμενο ως έχει μέσα στα πλαίσια αυτού του συμβιβασμού. Η κυρία Σπινέλη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για τις υποσχέσεις συνεργασίας, αλλά η στρατηγική ασφάλειας δεν με πείθει. Δηλαδή τι κάνει, εφαρμόζει την αρχή των ΙΠΑ για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Είναι κάτι σαν μία ε, Europol με πιο επεκτατικές δραστηριότητες. προβλέπει κατασταλτικά μέτρα αποκλειστικά. Δεν, γίνεται, δεν γίνονται τόσα πολλά για την ε, πρόληψη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρονται μόνο δύο φορές. Δυστυχώς καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα την τελευταία δεκαετία και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε περισσότερα νέα από την Αμερικανική Γερουσία για τα βασανιστήρια και για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω κατά πόσο το θέμα αυτό θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Κέλλερ για ένα λεπτό. ευχαριστώ πολύ εμείς οι πράσινοι Στηρίζουμε την ιδέα πως θα πρέπει να έχουμε στρατηγική την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί κόσμοι αισθάνονται ανασφαλείς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι μειονότητες, οι μουσουλμάνοι, οι μετανάστες οι οποίοι απειλούνται στη Γερμανία από τους φίλους όσων καθόνται προς τα δεξιά αυτής της αίθουσας καταπολέμηση του εγκλήματος που είναι για παράδειγμα η απάτη ή το εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος αλλά ξέρετε πως αυτή η τάση του να είναι όλοι ύποπτοι μας ανησυχεί. Δεν μπορούμε να τους υποπτευόμαστε όλους. Δεν είναι ο τρόπος αυτός για να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ελευθερίες μας. Αυτό άλλωστε επιδιώκουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε περιοριζοντάς τις. Και δεν πιστεύω πως θα έπρεπε να κλείσουμε τα σύνορά μας έτσι ώστε να κλείσουμε εκτός σύνορων κάποιους ε, εξτρεμιστές ε, που μας απειλούν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανοιχτή, να υποδέχεται και να καλωσορίζει όσου προέρχονται εκτός, από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρει ένα χώρο ασφάλειας αλλά και ελευθερίας στο εσωτερικό της. Αυτό είναι βασικό για μας. Ευχαριστώ κύριος Μποργέζιο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έναντι των μεγάλων απειλών, αρκεί να σκεφτούμε το Πακιστάν, πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική είναι πολύ αδύναμη και ανακριβής. Στα πιο σοβαρά σημεία δεν μας λέτε τι ακριβώς θα κάνετε. Τι θα κάνετε στην περίπτωση ας πούμε των σκοπευτών, των ελεύθερων σκοπευτών όπως είδαμε και στην περίπτωση του Πακιστάν. Επίσης, τι θα κάνετε με τους ξένους ε, μαχητές που επανέρχονται στη χώρα τους, δηλαδή αυτοί οι κύριοι οι οποίοι γίνονται τρομοκράτες και επανέρχονται στη Βιέννη, στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και τρομοκρατούν, προβάλλουν την τρομοκρατία. Τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να τους ιχνηλατήσετε και να μην μπορούν να επανέλθουν. Αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια μας. Επίσης, τι θα γίνει με τους ε, παράνομους. Με το Mare Nostrum στην ουσία τι κάναν, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 150.000 πανφτωχοί άνθρωποι. Δεν μας λέτε τι ακριβώς θα γίνει στο μέλλον. Κύριε Ντέλα Βέντοβα, δεν μας απαντήσατε τι θα κάνετε γιατί το ίμιση των παράνομων προσφύγων στην ουσία δεν έχουν ταυτιστεί, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, κυκλοφορούν στην Ευρώπη ανάμεσά μας. Πολύ ωραία ασφάλεια. Κύριε Μποργέζιο, έχετε μία γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ισδεχόφσκι. Την δέχεστε? Κύριε Ισδεχόφσκι, έχετε μισό λεπτό να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε πώς σκοπεύετε να αποτρέψετε αυτούς τους ε, μοναχικούς ε, ε, που μπορεί να διαπράξουν βία εγκλήματα αυτούς τους σκοπευτές που αναφέρατε ή τους μοναχικούς λύκους. Κύριε Μποργέζο, έχετε το λόγο, μα είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που δεν κάνουμε ας κλείσουμε τα Ισλαμικά κέντρα ε, εκεί όπου δυστυχώς οι Ισλαμιστές λαμβάνουν εκπαίδευση μίσους. Υπάρχουν βεβαίως πολλά τζαμιά που δεν γίνεται αυτή η εκπαίδευση, αλλά και σε πολλά γίνεται, προετοιμάζονται αυτοί οι Ισλαμιστές ε, τρομοκράτες, ακόμα και αν είναι μοναχικά στοιχεία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα και δικαστικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα σπίτια μας. Αυτή ήταν η πολιτική μας, γιατί τους αφήσαμε να μπούμε στο εδάφι μας. Υπάρχει και άλλο, άλλη μια γαλάζια κάρτα από την κυρία Σπινέλη. Τη δέχεστε, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μποργέζιο αν θυμάται τι είναι το Mare το οποίο σταμάτησε. Δεν ήταν για την εισδοχή των προσφύγων αποκλειστικά. Ήταν ένα σχέδιο για να σώσουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν να βαγήσει για να βρεθούμε εκεί που πνίγονταν και να τους βοηθήσουμε. Ναι βεβαίως, έχει δίκιο κυρία Σπινέλη. Αυτό ήταν ο αρχικός στόχος όμως δυστυχώς η δράση ήταν καταστροφική γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχαν και πολλοί ενδυνάμοι τρομοκράτες, γιατί φυσικά υπάρχει το δικαίωμα του ασύλου, της χορήγησης ασύλου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μπουν στο έδαφος μας και γιατί δεν υπήρχε φωτοαναγνώριση έτσι ώστε να είμαστε κάπως πιο ήσυχοι. Η κυρία Βόιζενμπεργκ για 1,5 λεπτό. Επίτροπε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνθήκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει να δούμε τα καινούρια δεδομένα. Ποια είναι αυτά. Είναι το διασυνοριακό έγκλημα το διεθνές έγκλημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι εγκληματικές οργανώσεις που αφορούν σε εμπόριο ανθρώπων εμπόριο οργάνων εμπόριο ναρκωτικών εμπόριο λευκής αρκός κυρίως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και γενικά απάτες και εγκλήματα τα οποία δεν είχαν ποτέ αυτή τη διάσταση η δεύτερη παράμετρος είναι η τρομοκρατία με καινούρια δεδομένα με θρησκευτικά κίνητρα και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανεστάλλει η εφαρμογή της οδηγίας που αφορά στη διατήρηση δεδομένων δυσχεραίνει τον κυρίαρχο τομέα που αφορά στην κουλτούρα της ευρώπης σε αυτό που αναφερθήκατε κύριε επίτροπε στην πρόληψη. απαιτείται λοιπόν μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία σε ολιστική μορφή θα μπορεί να συγκεράσει τις αντίθετες απόψεις που διατυπώνονται στις νομοθεσίες των κρατών μελών μια νομοθεσία η οποία θα διαπνέεται από τις αρχές της ενότητας της αναλογικότητας της αλληλεγγύης και κυρίως της δικαιοσύνης. μόνο έτσι μπορεί να αποτροπεί το φαινόμενο και μόνο μπορεί έτσι να συνεργαστούν οι θεσμοί η αστυνομία η δικαιοσύνη για την καταστολή ενός φαινομένου η πρόληψη του οποίου δεν μπορεί να το αποτρέψει. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάιντεν για ένα Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όλοι έχουν δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς και να ζουν ελεύθεροι από φόβο. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συζήτηση. Βέβαια, την ασφάλεια δεν μπορούμε να την εξασφαλίσουμε περιορίζοντας την ελευθερία. Πρέπει να υπάρχουν διάφορες και αμοιβαίες σχέσεις με την από, από την αποτελεσματική βεβαίως καταπολέμηση της τρομοκρατίας για την οποία χρειάζεται η Ευρώπη μια κοινή στρατηγική, μια κοινή πολιτική για την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Από την προηγούμενη θητεία ε, είχαμε κάποιες ε, σημαντικές βελτιώσεις. Για να εξασφαλιστεί όμως πάνω απ' όλα η ασφάλεια χρειάζονται συνθήκες πλαισίου, η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου η οποία υπάρχει μόνο όταν λειτουργούν οι θεσμοί που επιβάλλουν το σεβασμό του νόμου και του δικαίου, όπου υπάρχει η κοινωνική ασφάλιση, ασφάλεια επίσης. Όπου χάνεται η κοινωνική ασφάλεια, τότε η ανασφάλεια μέχρι και η εγκληματικότητα έρχονται γρήγορα. Η πολιτική ασφάλεια λοιπόν πρέπει με αυτή την έννοια να θεωρηθεί ολιστικά δηλαδή. Ιδάλλως με, την, ε, ε, με πιο αυστηρούς ελέγχους. Δεν μπορούμε παρά μόνο να ασκήσουμε περισσότερες πιέσεις και προβλήματα δεν πρόκειται να λύσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η κατάσταση ομοιρίας ε, όπου κρατήθηκαν τόσοι αθώοι στο Σίδνεϊ από έναν Ισλαμιστή μας φέρνει μπροστά στην πραγματικότητα. Μας ανοίγει τα μάτια. Δεν πρέπει να διερωτώμεθα εάν πρόκειται κάτι τέτοιο να ξανασυμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πότε στο Άμστερνταμ θα είναι, στο Βερολίνο θα είναι κάποιο Ισλαμιστή και δεν θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν, οι μαχητέ Ισλαμιστέ, τζιχαντιστέ. Ε, δεν αναγνωρίζουμε διαρθρωτικά τους, τομείς, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, δεν τους αναγνωρίζει η πολιτική το σχέδιο αυτό, είναι μια παροδία. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα πόσοι τζιχαντιστές έφυγαν για να πολεμήσουν για το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Πόσοι από αυτούς γύρισαν πίσω σε ευρωπαϊκά εδάφη. Πότε θα αναγνωρίσετε το Ισλάμ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ασφάλειά μας. Και για να ολοκληρώσω. Η ασφάλεια είναι εθνικό ζήτημα. Όσο όμως δεν το αντιλαμβάνονται αυτό οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν θα δοθούν απαντήσεις. Η λύση είναι πιο πολύ έλεγχη, η αφαίρεση των διαβατηρίων από αυτούς τους τσιχανιστές ώστε να μην μπορούν ποτέ να γυρίσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η κυρία Μετσόλα, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν πάρα πολύ για το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας. Οι πρόσφατες, ε, τα πρόσφατα γεγονότα, ιδιαίτερα του Πακιστάν, είναι τρομακτικά και αποτροπιαστικά. Δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσω τη φρίκη που αισθάνθηκα όταν διάβασα ότι παιδιά που είχαν πάει στο σχολείο τους έχασαν τη ζωή τους από το χέρι τζιχαντιστών. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των συνόρων με εσωτερική και εξωτερική διάσταση ε, μια στρατηγική η οποία θα πρέπει την ε, ε, λαθρεμπορία ανθρώπων να την θέσει σε κύρια προτεραιότητα να χτυπήσει τα κέρδη αυτών των οργανωμένων εγκληματιών που είναι το, ο, ο κύριος στόχος μας και η πιο αποτελεσματική δράση και αυτοί οι μαχητές, οι, Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι δηλαδή πολίτες οι οποίοι πάνε να πολεμήσουν για την Τσιχάτη για να γυρίσουν μετά στην Ευρώπη πρέπει να πληγούν αποφασιστικά. Και αναφέρομαι και στη Λιβύη, γιατί εμείς στη Μάλτα ζούμε από πολύ κοντά το χάος που επικρατεί στη χώρα αυτή. Επικρατεί χάος και ήδη ο συντονιστή που έχουμε στη χώρα μα για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση τρομοκρατία ήδη προειδοποιεί πω επεκτείνεται το ΙΚΙΛ, το Ισλαμικό κράτο Ιράκ και Λεβάντε, και στη Λιβύη. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ασφάλεια και θεμελιωδών ελευθεριών, αλλά να είμαστε πάνω απ' όλα προετοιμασμένοι για του κινδύνου που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μια στρατηγική η οποία δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιώτοβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ασφάλειας μέσω μίας ασφαλούς στρατηγικής. Χρειάζεται μία πιο αποτελεσματική ασφάλεια, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες και δυσίωνες απειλές. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και τη διαφθορά. Το 2016 η Επιτροπή θα υποβάλει μια νέα έκθεση κατά της διαφθοράς. Χρειάζονται όμως μέτρα για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του σφετερισμού δημοσίου χρήματος πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε ε, να αντιμετωπίσουμε πολλές απειλές. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί το 2010 ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ξένους ε, μαχητές πρόταση της αστυνομίας συνόρων ήταν κάτι το οποίο ήταν το πολύ μακρινό. Τώρα όμως βλέπουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να ενισχυθεί και η Frontex στα σύνορα μεταξύ ε, Βουλγαρίας ε, και Τουρκίας, η Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενίσχυση της Frontex είναι ένα από τα μέτρα. Η στρατηγική εσωτερική ασφάλειας έχει αποδειχθεί γενικά επιτυχής και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ανανεωθεί. Να ανανεωθεί. Δυστυχώς όμως οι προτινόμενοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί η απειλή κατά της Ευρώπης περισσότερο θεραπεύουν ε, παρά προλαμβάνουν ένα κίνδυνο. Θα εξηγήσω τι εννοώ είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στις χώρες της ε, νοτιού ευρώπης σειραίουν εκατοντάδες χιλιάδες παρανόμων μεταναστών. από την εμπειρία που έχω από την πατρίδα μου την ελλάδα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από τα διεθνή κυκλώματα ως μέσον για να υλοποιηθούν τέσσερις από τις μεγαλύτερες απειλές κατά της ευρώπης τις οποίες φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας. οι απειλές αυτές είναι το εμπόριο ανθρώπων το εμπόριο παραποιημένων αγαθών η διακίνηση ναρκωτικών και η τρομοκρατία και αν μου πείτε ότι είμαι υπερβολικό επειδή στα ανατολικά σύνορα τη ελλάδο μαζί με τι εθνικέ δυνάμει ασφαλεία συνεργάζονται και οι δυνάμει τη frontex θα σα πω ότι αυτό δεν είναι σωστό διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ταξιδιώτε οι οποίοι ταξιδεύουν ω τουρίστε στην ευρώπη. άρα η απλή καταγραφή του δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. αν θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη δομή ε, στρατιωτική εσωτερική ασφαλεία θα πρέπει να περιλάβει αυτή και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζεται από του παράνομου μετανάστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόνη για 1,5 λεπτό. Η νέα εσωτερική στρατηγική ασφαλείας είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε τις μεταλλασσόμενες απειλές. Ε, έγκλημα, κύβερνο έγκλημα, κυβερνοτρομοκρατία. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογίες, νέα νομοθεσία, νέο είδος συνεργασίας μεταξύ χωρών. Για παράδειγμα, η οδηγία για, τα, ε, για την ασφάλεια των δικτύων. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την οικονομική και οργανωτική δυνατότητα που έχουν οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Δεν θα πρέπει απλώς να, κάνουμε μια, να δίνουμε μια απόκριση στα όσα συμβαίνουν. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν την ε, νέα τεχνολογία για τους δικούς τους στόχους και online μπορούν ως εγκληματικές οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν πάρα πολλές υπηρεσίες. Πολύ δύσκολα μπορεί να εντοπίσει κανείς τέτοιου είδους έγκλημα και οι απώλειες ε, για την διεθνή οικονομία είναι ετησίως γύρω στα 250 δις. Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο τρόπος που σχεδιάζουμε την ασφάλειά μας και να έχουμε λύσεις που θα εισάγουμε ε, μαζί με νέα προϊόντα και νέες στρατηγικές. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται οι ιδιοκτικές αρχές να συνεργαστούν με τους ακαδημαϊκούς κύκλους, με τους επιχειρηματικούς κύκλους, όπως επίσης και με τους ε, ερευνητές. Πρέπει όμως να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας αφενός και θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτούν. Αυτό θα αποτελέσει την ε, ακρονία λίθο της νέας πολιτικής. Στο παρελθόν είπαμε χρειάζεται συνέπεια στην προσέγγιση που ακολουθούμε για να εξασφαλίσουμε την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Άρα λοιπόν συνεργασία με τους εταίρους μας, με τρίτες χώρες. Αυτό είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Ο κύριος Μπέκερ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πετροπέ, και κύριοι συνάδελφοι. Το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε αύριο της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών για την τραγωδία της Λαμπεντούζα κλείνει, έχει περάσει ένας χρόνος. Ε, νομίζω θα πρέπει να αποτελέσει το μύτο της Αριάδνης για την ε, Επιτροπή. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω την Επιτροπή να συνεχίσει ακόμη περισσότερο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου των παράνομων μεταναστών Άρα χρειάζονται checkpoints, σημεία ελέγχου στα τρίτα κράτη που πρέπει να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε ελάχιστα, ελάχιστες ποσοστώσεις για υποδοχή μεταναστών για όλα τα κράτη, με κυρώσεις αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Θέλουμε επίσης εντατικό και εντεταμένο έλεγχο κατά των διακινητών, του λαθρεμπορίου ανθρώπων με τη συνδρομή βεβαίως της Frontex και τρίτων έχουμε μια αύξηση του προϋπολογισμού για τη Frontex που θα ψηφιστεί αύριο ευτυχώς. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει επίσης διατυπώσει προτάσεις για την εσωτερική ασφάλεια που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εάν αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη, εάν υλοποιούνται, μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Και αυτός είναι ο δρόμος που προτείνω στην Επιτροπή. Ο επόμενος ομιλητής για ένα μισή λεπτό, ο κύριος Τσεκόφσκι. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και θετική έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ελευθερία των πολιτών. Αυτό είναι βαρισίμαντο έργο, όμως δεν θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με ένα τέρας νέων μέτρων που κανείς δεν θα μπορέσει να ελέγξει. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τα προϋπάρχοντα μέσα της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και να τα χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της ανανέωσης. Το θέμα της ασφάλειας προσλαμβάνει νέες διαστάσεις, όχι μόνο λόγω των σειράξεων σε όμορες περιοχές, αλλά επειδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπλώνεται η τρομοκρατία σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 3.000 Ευρωπαίοι συμμετέχουν σε διεθνείς σειράξεις. Μα πώς βρίσκονται εκεί. Θα πρέπει να σπάσουμε αυτό το δίκτυο που προσλαμβάνει νέα πρόσωπα για να πολεμήσουν σε άλλες χώρες. Αυτό είναι προτεραιότητα για όλους, πιστεύω. Μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye ένας ζητάει το λόγο, ο κύριος Τζαμπάτσκι, ο οποίος έχει και το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κυρίε και κύριοι συναδελφοί, διάβασα με προσοχή την έκθεση για την υλοποίηση της εσωτερικής πολιτικής ασφάλειας 2010-2014. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση μόνο θετική. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω κάποιε προσθήκε που μπορεί να βελτιώσουν την έκθεση και τι δραστηριότητε. Θα πρέπει να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία κατά τη διακίνηση. γιατί πέρα τη διακίνηση των ναρκωτικών υπάρχει όλο και περισσότερη διακίνηση ανθρώπων, λαθρεμπόριο ανθρώπων που προορίζονται να γίνουν πρωτοφολάδες ή ε, επέτες. Επίσης πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση. Πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο ο συσχετισμός μεταξύ του σλαμιστικού στοιχείου και του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια που αποτελούν σαφή απειλή για τους πολίτες της Ευρώπης. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Έχει το λόγο κύριε Αβραμόπουλε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα ελέγξαν πριν από λίγο από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έλεγα ότι ξεκινώ από μια βασική παρατήρηση. Ότι σε γενικές γραμμές όλοι συμφωνούμε ότι η ασφάλεια σήμερα είναι μία από τις βασικότερες προτεραιότητες όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνο όμως που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η συζήτηση αυτή και η πρωτοβουλία που αναλάβαμε να υιοθετήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή και για την ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. νέες μορφές απειλής για την ασφάλεια η οποία και αυτή είναι θεμελιώδε δικαίωμα και προστατεύεται από τη δημοκρατία από το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις κατακτήσεις του πολιτισμένου κόσμου από το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ευρώπη έχει στηριχθεί σε αυτές τις αρχές. το ότι δεν υπήρξε μια ολοκληρωμένη συνεκτική πολιτική ασφάλειας αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλες ήταν οι μορφές απειλής στο παρελθόν και άλλες τώρα. όπως λέει πρωτήτερα έχουμε την απροκάλυπτη απειλή της τρομοκρατίας η οποία δεν ξέρουμε πότε και πού θα χτυπήσει. το ζούμε δε αυτές τις μέρες. το οργανωμένο έγκλημα τους διακινητές και τους εμπόρους ανθρώπων τα κυκλώματα τους εμπόρους ναρκωτικών όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σε κάποιες γωνιές του κόσμου όπου το οργανωμένο έγκλημα έχει δέσει με την τρομοκρατία και τα οργανωμένα κράτη παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μέσα και δυνατότητες δεν έχουν καταφέρει να πατάξουν αυτό το φαινόμενο. προστατεύεται λοιπόν από αυτήν την ατζέντα εσωτερικής ασφάλειας ένα εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων που με μεγάλες θυσίες έχει κατακτήσει η ευρώπη και ο ελεύθερος κόσμος. θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμα φορά η πολιτική που φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να οδηγήσει την ευρώπη σε απομονωτισμό. το έχω πει χαρακτηριστικά δεν θέλουμε μια ευρώπη φρούριο. η ευρώπη πρέπει να είναι ανοιχτή. δεν πρέπει επίσης να συνδυάζουμε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία διότι αυτή η αντίληψη στο παρελθόν οδήγησε σε λάθος πολιτικές πάρα πολλές φορές και θυμίζω και μια ακόμα φορά σε αυτή την αίθουσα ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο προερχόμαστε από έθνη μεταναστών. γι' αυτό θα πρέπει όλη η προσέγγιση να γίνεται με εντελώς διαφορετικά κριτήρια. δεν μας λείπει όμως ούτε η τόλμη ούτε η αποφασιστικότητα. άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα είπατε και θα τα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη για την ε, κατάρτιση της τελικής μας πρότασης. θα ακολουθήσουν πολλές συζητήσεις και είμαι βέβαιος ότι μέσα από τον χώρο θα προκύψει ίσως μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές που θα διασφαλίσουν την ειρήνη τη σιγουριά την ασφάλεια την ελεύθερη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους λαούς της ευρώπης και μέσα από αυτό το μήνυμα η ευρώπη θα είναι πρωτοπόρος και σε ολόκληρο τον κόσμο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και κάθε μορφής απειλής που έχει σαν σκοπό να δυναμητήσει τα θεμέλια της παγκόσμιας δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα ο κύριος Δηλαβέντοβα να λάβει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντάχει, αγαπητοί βουλευτές, το Συμβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη το θέμα, προσδίδει μεγάλη σημασία στη γνώμη του Κοινοβουλίου και λάβαμε υπόψη και την επιχειρηματολογία σας. Θεωρούμε ότι η στρατηγική της εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να ανανεωθεί άρδιν και να προστατεύσει πλήρως τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη και τις ελευθερίες τους. Θεωρούμε ότι η ανανεωμένη στρατηγική θα πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας πριν δημιουργήσουμε νέα, μέσα στα πλαίσια μιας ολιστικής και εξισορροπημένης προσέγγισης, όπως ορίζουν οι συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να ε,